Uh, koleżanki i koledzy, ladies and gentlemen, please take your seats. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζουμε σε ένα λεπτό. Ε,